Good morning, everyone. Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Please be. Καλή σας μέρα, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καθίστε. Ας ξεκινήσουμε την σημερινή μας συνεδρίαση. Καλώς ήρθατε. Περνάμε στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης, ηλεκτρονική ψηφοφορία για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό έτος 2020 όλα τα τμήματα. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία θα δώσω το λόγο στον ε, κύριο Γκάλερ που είναι ο εισηγητής. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Προσοχή, θα μιλήσω γερμανικά. Θέλω να μιλήσω γερμανικά κατά εξαίρεση σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θέρμα για την εξαιρετική συνεργασία που είχε ως αποτέλεσμα ότι συνελικά καταλήξαμε σε 10 συμβιβαστικές που μπορέσαμε, μπορέσαν να μας βρουν σύμφωνους και προσδοκώ να έχουμε καλύτερη περαιτέρω συνεργασία. Ένα πράγμα που έκανε εντύπωση. Έχουμε πολλούς νέους συναδέλφους και πολλοί έχουν πολύ καλά επιχειρήματα και καλές προθέσεις. Θα ήθελα να εστιαστώ σε δύο ωστόσο τροπολογίες ε, που εγώ ε, πέριψα. Πρόκειται για τις 51 ε, και 56 αφορούν το gender-based violence και το legal abortion. Εγώ δεν είμαι κατά του να ασχοληθούμε με αυτά. Το κάνουμε ούτως ή άλλως ως Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη. Ωστόσο, Αυτές οι γενικές διατυπώσεις Use of EU funds uh, to support the rights around the world to access αυτά, αυτές οι γενικές διατυπώσεις δεν οδηγούν, uh, δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική τέτοιου είδους uh, σε ένα προπολογισμό όταν, υπάρχει, όταν έχουμε ένα κρατικό πρόγραμμα, ένα θεματικό πρόγραμμα ε, δεν λέμε θέλω περισσότερα λεφτά, λιγότερα λεφτά ε, θέλω τα ίδια, την ίδια χρηματοδότηση. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι θα μπορούσαμε να έχουμε μια γνωμοδότηση για ένα πρόγραμμα εκεί να συμπεριλάβουμε αυτές τις πληροφορίες αλλά όχι σε, στον προϋπολογισμό σε μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για τον προϋπολογισμό θέλω να αποφύγω να το στολίσουμε υπερβολικά να το κάνουμε σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο θα μπορούσε μια τέτοια τροπολογία να βάλει κανείς οποιαδήποτε άλλη ε, επιτροπή των γυναικών, των ε, ε, δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε θέλω να ξέρετε ότι παρότι είμαι διαθέσιμος φυσικά και είμαι σύμφωνος να ακολουθούμε αυτές τις πολιτικές σε όλες τις χώρες, δεν προσθέτει καμία αξία σε, να κάνουμε μια να προσθέσουμε αυτό σε κάποια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Προπολογισμών, ούτε εδώ Οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω και την κατανόησή σας. Ε, ε, εγώ δεν δέχομαι αυτές τις δύο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαι κατά. Για τις 51 και 56 λοιπόν ε, ήθελα απλά να καταστήσω αυτό σαφές ότι εδώ έχουμε μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για τον προπολογισμό και όχι κάτι στο οποίο θα αναφέρουμε τα πάντα και που θα πρέπει να προλαμβάνει όλε τι πτυχέ για όλα τα θέματα. Αυτά ήθελα να πω στην αρχή τη θητείας γιατί βρισκόμαστε και σε μια διαδικασία προπολογισμού για πρώτη φορά και ό,τι θεωρεί κανεί ε, σωστό φυσικά πρέπει να το περιλαμβάνει και στον προπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλερ. Υπάρχει κάποιο άλλο που θα ήθελε το λόγο, κύριε Νόημαν. Πρέπει να πω ε, προσοχή γερμανικά. Είμαι λίγο έκπληκτη. Ε, αυτά τα θέματα ανήκουν και σε αυτό το τομέα, οπότε πρέπει να τα τονίσουμε. Ε, σε εποχές όπως σήμερα όπου υπάρχει το θέμα των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ και ε, τη ισότητα των φύλων, πρέπει να πούμε ότι κομμάτι τη εξωτερική μα πολιτική περιλαμβάνει και αυτά στον προπολογισμό. Θέλουμε να δείξουμε ότι με τον προπολογισμό μας de facto ασχολούμαστε και με αυτά τα θέματα. Ε, στον επόμενο προπολογισμό θέλουμε να μιλήσουμε για gender mainstreaming. Αυτό είναι σημαντικό πολιτικά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπιωτικόφερ, παρακαλώ. Έχω μια ερώτηση προς τον Μιχαήλ Γκάλερ. Σε αυτή την ε, θητεία, κύριε Γκάλερ, πώς θα ξέρουμε πότε το όχι το δικό σας σημαίνει ότι είστε υπέρ. Όταν έχω ένα πρόγραμμα που αφορά μια συγκεκριμένη χώρα ή ένα συγκεκριμένο θεματικό τομέα, όπου μπορώ αντικειμενικά να συμπεριλάβω το θέμα, τότε θα μιλάω υπέρ αλλά μιλάμε πολύ συγκεκριμένα για μια χώρα ή για μια, ένα συγκεκριμένο εγχείρημα ε, ε, για το οποίο προσπαθούμε, αλλά όπως είπα, σε μια γενική γνωμοδότηση για τον προπολογισμό της Επιτροπής μας Εξωτερικών Υποθέσεων, θεωρώ ότι τέτοια θέματα δεν μπορούν να συμπεριληφθούν. Διότι τι να κάνει με αυτά η Επιτροπή Προπολογισμών. Δεν τις χρησιμεύουν σε τίποτα. Κάνουμε την πολιτική, ναι, αλλά πολύ συγκεκριμένα στη χώρα Α, Γ, όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι προπολογισμοί που προβλέπονται και εκεί είναι μια χαρά. Αλλά εδώ, ε, σε μια γενική γνωμοδότηση, να λέμε τέτοια ε, γενικόλογα πράγματα, κατά την άποψή μου δεν είναι σωστό και ε, δεν θέλουμε να δώσουμε κακή φήμη στην Επιτροπή μας από την αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ως πρόεδρος λοιπόν θα έλεγα σιγά σιγά να περνάμε στο ψηφοφορία να μην κάνουμε εκτενή συζητήσει αυτή τη στιγμή. Δίνω σε δύο ακόμα το λόγο και μετά μπορούμε να το κλείσουμε. Κυρία Φωνβίζε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Φανόημαν πήρε ακριβώ τα λόγια από το στόμα μου. Συμφωνώ απόλυτα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ψηφίσετε υπέρ της τροπολογίας 51. I just have Διαφωνώ με τον κύριο Γκάλερ. Θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβει τα, τους αριθμούς των τροπολογιών που θέλει να ψηφίσουμε κατά. Ο κύριος Γκάλερ, 51 και 56 είναι οι τροπολογίες. Ο κύριος Γκάλερ ζητά από τους συναδέλφους που υπέβαλαν τις τροπολογίες 51 και 56 να τις αποσύρουν. Το δέχονται, φαντάζομαι όχι βέβαια. Όχι. Οι άλλοι δύο οι άλλοι τρει, όχι. Ούτε. Ο κ. Γκάλερ ήταν σαφή, Α περάσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά εποχέ, απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά Εποχέ. απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 2 υπέρ κατά Εποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά Εποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά Εποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Εποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Εποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Εποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Εποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Εποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονική επιβεβαίωση για την 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 27 κατά, 24 υπέρ. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αλλά ελέγχουμε ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, Τι γίνεται τώρα. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμό 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Όχι, εγκρίνεται, συγγνώμη. 37 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 38 και 39 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λείπει μία ψήφος. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. «35 κατά 19 υπέρ» ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί δεν το, γιατί δεν το βάλαμε στην οθόνη, γιατί δεν το αναρτήσαμε. Συμβαίνουν αυτά. 42 της κύριος Φωτίγα. Υπέρ. Τη 40, ε. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Καστάλτο, 40. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Ε, ηλεκτρονική επαλήθευση. Αυτή τη φορά βάλτε το και στο βίντεο το αποτέλεσμα. Λήξη ψηφοφορίας. Σαράντα ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Για τη 42 άρχεται η ψηφοφορία. Λείπει μία ψήφος. Ωραία. Κλείνουμε. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Εποχέ εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Εποχέ απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Εποχέ εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. εποχέ. απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές Επαλήθευση, ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Λείπει μία ψήφος. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Καινούρια παράδοση αυτή τα χειροκροτήματα μετά ουσιοφορίας. Ανοιχτό είμαι σε αλλαγέ, αλλά είναι πολύ πρωτότυπο έτσι, και ενοφανέ. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Έναρξη τη ψηφοφορία. Λήξη της πληροφορία, εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές. 62 ελέγχεται, ηλεκτρο... Ε, επαληθεύεται ηλεκτρονικά. Ένα αξίσου ψηφοφορίας. Λήξη. Απορρίπτεται. Με 12 αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά στο σύνολο της νομοδότησης όπως τροποποιήθηκε έναξης πληροφορίας. Δύο, μία ψήφος λείπει. Τελευταία σας ευκαιρία. Λήξη της πληροφορίας. Εγκρίνεται 42 υπέρ 12 κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Φτάνουμε στη λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Fine. So we come to the end of the electronic vote. Οι Αυστραλοί φίλοι μας βρίσκονται ήδη παρόντες στην... Έχουν φτάσει, Ρακέλ. Σε δύο λεπτάκια θα είναι εδώ. Παρακαλώ πολύ, κρατήστε τις θέσεις σας. Σε, α, σε πέντε λεπτάκια λέει η Ρακέλ. Ωραία, συνεχίζουμε ξανά σε πέντε λεπτά. Είναι κάποιος από τη γραμματεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων που παραμένει στην αίθουσα. Μήπως έχετε κάποιο νέα, κάποιες εξελίξεις. Μας είπατε ότι σε πέντε λεπτά θα έρθουν οι Αυστραλοί φίλοι μας. Μήπως ε, πέντε λεπτά στην Αυστραλιανή Ήπειρο ε, έχει, είναι διαφορετικός χρόνος που μετρέται διαφορετικά. Αναρωτιέμαι. Δεν καταλαβαίνω μήπως ε, Πώς είναι δυνατόν να καθυστερούν παραπάνω από 5 λεπτά. Our guests are already in the building. Μήπως έμπλεξαν με τη βελγική αστυνομία. Α, είναι ήδη στο κτίριο. Από ό,τι μαθαίνω. Probably hidden Μήπως κρύφτηκαν κάπου. Συνάδελφοι, επειδή έχουμε καθυστερήσει, θα ήθελα ευθύ αμέσω να συνεχίσουμε την πρωινή μας συνεδρίαση. Έχουν φτάσει οι προσκεκλημένοι μας από την Αυστραλία. Θα ήθελα να καλωσορίσω επισήμως τον αξιότιμο Κέβιν Άντριου, τον αρχαιότερο βουλευτή στην Βουλή των Αντιπροσώπων της Αυστραλίας. Φαντάζομαι ε, σας προκαλεί περιπέργεια η λέξη, γιατί στα αγγλικά αυτό το ονομάζουμε father, ο πατέρας δηλαδή ε, του ε, οίκου των αντιπροσώπων της Αυστραλίας. Καλωσορίσω την κυρία Τζοάν Ριάν, την αρχηγό της κοινοβουλευτικής ομάδας στην Βουλή των Αντιπροσώπων της ε, Αυστραλίας, τον αξιότιμο Ντέμιαν Ντραμ, μέλος της μόνιμης σταθερής κοινή επιτροπής για εξωτερικές υποθέσεις άμυνα και εμπόριο του Αυστραλιανού Κοινοβουλίου και τον γερουσιαστή αξιότιμο Τζέιμς Μαγκράθ. Δεν έχουμε ναι. καθώς και την ε, γερουσιαστή Πολίνη Χάνσον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αυστραλία έχουν πολύ μακριά, μακρόχρονες διπλωματικές σχέσεις. Από το 1962 η δική μας αντιπροσωπεία άρχισε να λειτουργεί επισήμως στην Αυστραλία το 1981. Θα ήθελα ε, να κάνω λίγα σχόλια πριν ε, προβούμε στην ανταλλαγή απόψεων. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αυστραλία είμαστε εταίροι που έχουμε την ίδια νοοτροπία και έχουμε και το ίδιο όραμα και την ίδια άποψη για διάφορα θέματα και για την εξωτερική πολιτική, όπω είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κλιματική αλλαγή, η έρευνα, η καινοτομία, η καταπολέμηση τη τρομοκρατία και η ανάγκη να παραμείνει η παγκόσμια τάξη πραγμάτων με βάση το κράτο δικαίου, με βάση το δίκαιο και την πολυμέρεια. Αυτή η σχέση ενισχύθηκε ε, διότι μπήκαμε σε μια νέα περίοδο στρατηγική συνεργασία με την ολοκλήρωση τη συμφωνία Πλαίσιο το 2017 μεταξύ ε ΕΕ και Αυστραλίας, την οποία προσυπέγραψε και ενίσχυσε το Κοινοβούλιο το 2018. Ε, τώρα, στη νέα κοινοβουλευτική μα θητεία, θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο εμπόριο. Γίνονται διαπραγματεύσει για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Αυστραλία. Εμεί στηρίζουμε τι διαπραγματεύσει για μια τέτοιου είδου συμφωνία φιλόδοξη και συνολική, που να περιλαμβάνει όλα τα θέματα. Χρειάζεται να ε, συνεργαστούμε για να έχουμε μια κοινή πλατφόρμα για να επιδιώξουμε τα, μας, τα κοινά μας συμφέροντα, να ανταλλάξουμε ιδέες και πληροφορίες. Νομίζω ότι η κοινοβουλευτική διπλωματία εξελίσσεται και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους Αυστραλιανούς συναδέλφους και να δώσω το λόγο στον αξιότιμο πατέρα ε, του ε, Κοινοβουλίου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αυστραλίας. Αυτό είναι ο επίσημος όρος σας, ίσως θα έπρεπε να τον εξηγήσετε. Καλώς όρισατε και πάλι, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τα θερμά σας λόγια, για την πολύ θερμή σας υποδοχή. Πριν έρθω στον όρο ο πατέρας ε, του Κοινοβουλίου, να σας πω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά για εμάς, για την αντιπροσωπεία μας που είμαστε εδώ στις Βρυξέλλες. Σήμερα το πρωί αργότερα, θα έχουμε την επίσημη ε, συνεδρίαση που θα ε, τιμά τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοβουλίων τα τελευταία 40 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και η σχέση των δύο οίκων των αντιπροσώπων θα γίνει όλο και πιο ε, στενή τα επόμενα χρόνια. Και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό καθώς και στην ε, Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας. Εγώ εξελέγη το 1991 όρος πατέρας του οίκου των αντιπροσώπων χρησιμοποιείται για να σηματοδοτήσει τον αρχαιότερο. Εγώ δεν το νιώθω βέβαια αυτό ότι είμαι αρχαιρότερό και δεν θέλω καθόλου και να με θεωρήσετε και παππού. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι μεγάλη μου τιμή που εκλέγομαι από το 1991 και είμαι το αρχαιότερο μέλος της Βουλής μας. Υπάρχουν δυσκολίες και όντω τι βιώνει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Εμείς ε, θεωρούμε όμως ότι η σχέση μας με την Ευρώπη είναι εξαιρετικά ισχυρές και θέλουμε να ενισχυθούν έτσι περαιτέρω στο μέλλον. Παρόλο που η σχέση μεταξύ Ευρώπης και Βρετανίας από ό,τι φαίνεται φτάνει στο τέλος της και εμείς δεν έχουμε ιδιαίτερες απόψεις γι' αυτό, αυτό είναι θέμα ευρωπαϊκό. Σε κάθε περίπτωση, από πλευράς εμπορικής, με ή ε, εκτός τη Βρετανία, η Ευρώπη παραμένει ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός μας εταίρος στον κόσμο. Και θέλω να το πω αυτό, διότι ανεξαρτήτως του ιστορικού υποβάθρου μας και της ιστορικής μας διαδρομής κοντά ε, στη Βρετανία, ε, το γεγονός που παραμένει ότι η Αυστραλία έχει σύνδεση με την Ευρώπη η οποία ξεπερνά τα βρετανικά σύνορα και το βρετανικό πλαίσιο. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά είχαμε δεχθεί μεγάλη μετανάστευση από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Στην εκλογική μου περιφέρεια έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό που κατάγεται από την Ελλάδα, από την Ιταλία ή από αλλού. Και είναι πολύ θερμέ και στενέ οι σχέσει μα με πάρα πολλέ ε, περιοχέ στην Ευρώπη και θα συνεχίσουμε να καλλιεργούμε αυτέ τι σχέσει στο μέλλον. Άλλωστε, ε, ο Αυστραλιανό λαό είναι πρακτικό λαό και παρά του ιστορικού δεσμού. Δεν θα αφήσουμε να μας κυριαρχήσει η συναισθηματικότητα. Θέλουμε να έχουμε πολύ ισχυρές σχέσεις με την Ευρώπη, ούτε, όχι μόνο εμπορικά, αλλά και οικονομικά και πολιτισμικά. Και τα λόγια σας είναι πολύ σημαντικά, κύριε Πρόεδρε, προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και από πλευράς ασφαλείας. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή αγοράζουμε στρατιωτικό εξοπλισμό, όχι μόνο πλοία ε, και τεθωρακισμένα και αεροσκάφη, αλλά επειδή έχω θητεύσει στο Υπουργείο Αμήνη στην Αυστραλία, τα γνωρίζω και αγοράζουμε από ευρωπαϊκέ εταιρείε, από ευρωπαϊκέ χώρε. Είναι σχέση αυτή πολύ σημαντική, πολύ στενή, γιατί το θέμα τη ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να ε, συνεχίσουμε τη συνεργασία στο μέλλον, να δούμε πώ μπορούμε να ευημερίσουμε αμφότεροι λαοί προ όφελο των λαών τη Ευρώπη και προ όφελο του λαού τη Αυστραλία. Αυτό πρέπει να γίνει με κανόνε συγκεκριμένου, είτε πρόκειται για την οικονομία, είτε πρόκειται για τη στρατηγική μας τοποθέτηση. Σε κάθε περίπτωση η Αυστραλία, όπως και εσείς, πιστεύει σε ένα ισχυρό σύστημα ε, ρυθμίσεων, ε, κανονισμών ένα νομικό πλέγμα το οποίο μας καθιστά μέρος του σύγχρονου κόσμου και πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη θερμή σας υποδοχή. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για εμάς που βρισκόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ τον Κέβιν Άντριους για τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις. Μήπως κάποιος άλλος από τους Αυστραλιανούς συναδέλφους θα ήθελε να πει δύο λόγια. Ωραία μιλάει ο πατέρας εξ ονόματος όλων ημών. Μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις ε, και τη συνομιλία με τους προσκεκλημένους μας από την Ελέκτρη του Κόσμου και δίνω το λόγο ανάλογα με τις ομάδες. Ξεκινάμε με τον κύριο Ζικόσκη. Hello. Um, <clears throat> I'm glad you mentioned Καλημέρα σας. Χαίρομαι που αναφερθήκατε για την κοινή μα δέσμευση για το ελεύθερο εμπόριο. Ο γύρο τη Δόχα φυσικά απέτυχε, αλλά έρχεται το Brexit. Και οι Βρετανοί υπολογίζουν ότι θα έχουν μια φανταστική εμπορική συμφωνία με την Αυστραλία. Πόσο πιθανό το βλέπετε και πόσο γρήγορα μπορεί να τεθεί σε ισχύ το εμπόριο μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Αυστραλίας πόσο μπορεί να αναπτυχθεί για να αντισταθμίσει την απώλεια που θα έχει στο εμπόριο η Αγγλία με την ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Να, κάνουμε, να ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις. Ωραία. Ο, ε, ο συνάδελφος Χαβιενάτ. Ο κ. Νάρτ. Η πρώτη ερώτηση που είχα ήταν αυτή που έθεσε ο κ. Σικόρσκι. Έχω όμως και μια δεύτερη. Κίνα. Η Κίνα ε, είναι μια ισχυρή δύναμη η οποία μπλοκάρεται από τα νησιά που ξεκινούν στην Ιαπωνία και τελειώνουν στην Ταϊβάν ε, και συνεχίζονται και προς τις Φιλιππίνες. Οπότε η είναι μια γεωγραφική πραγματικότητα μαζί με μια άλλη που είναι η επέκταση στον ειρηνικό ε, της Αυστραλίας αυτή τη φορά γιατί και η Αυστραλία θα ήθελε να υπερβεί αυτές τις νήσους και να αναπτυχθεί στον ειρηνικό Παππούα, Νέα Γουινέα, Κυρίμπας και αλλού όπου η Αυστραλία θα ήθελε να έχει ε, μεγαλύτερη παρουσία αλλά να έχει πιο πολύ παρουσία η Κίνα ναυτικές βάσεις. Ε, η ασφάλεια λοιπόν της Αυστραλίας θα επηρεαστεί από, αυτές, από αυτές τις ετάσεις και προθέσεις της Κίνας να επεκταθεί στον Ειρηνικό ωκεανό με στρατιωτική παρουσία. Next is Berg. Συνάδελφος κύριος Μπέργκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω θερμά την Αυστραλιανή αντιπροσωπεία μας. Συνδέουν όχι μόνο ε, πολιτισμός και εμπόριο, αλλά και θέματα πολιτικής ασφαλείας. Θα ήθελα να απευθύνω τα εξή ερωτήματα, βασικά ζητήματα στα οποία εστιάζεται η Αυστραλία, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, ε, οι δραστηριότητες καταπολέμησης της τρομοκρατίας και ειδικότερα για την Ισλαμική τρομοκρατία. Ποια είναι τα βασικά σημεία που υποστηρίζει και η Αυστραλιανή κυβέρνηση. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Ο κύριος, ο κύριος Μπουτικόφερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίζω τους φίλους μας στην Αυστραλία. Ε, θα ήθελα να σχολιάσω το θέμα της συνδεσιμότητας. Ήδη την περασμένη Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε μια, ένα πολύ μεγάλο συνέδριο για τη σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ασίας. Η Αυστραλία ήταν παρούσα με πολύ μικρή αντιπροσωπεία ενδιαφέρεστε να προωθηθεί ένα τέτοιο ζήτημα σύνδεση, συνδεσιμότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ασία, συμπεριλαμβανομένη και τη Αυστραλία. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από 1,5 περίπου χρόνο δημοσίευσε κάποια συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και των χωρών Ασία και Ειρηνικού σε θέματα ασφαλείας. σε ποιο βαθμό η Αυστραλία έλαβε γνώση ε, και έλαβε υπόψη αυτά τα συμπεράσματα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ε, τρίτη ερώτηση. Στην, ε, στην, στην Αυστραλία γίνεται μια συζήτηση για το ρόλο της Κίνας. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι συνεξελίξη. Ευχαριστώ πολύ. Το ECR έχει το λόγο. Ο κύριος Τέρτς. Καλώς ήρθατε, Αυστραλοί φίλοι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την πολιτική μετανάστευση που ακολουθείτε, τη μεταναστευτική σας πολιτική η Αυστραλία βασίστηκε στην δημιουργία, κατά τη δημιουργία της στην μετανάστευση. Πέρασε μια κρίση πριν από κάποια χρόνια και ακολουθεί μια πολιτική εξήγησης της χώρες προέλευσης ε, που είχε φαίνεται πολύ καλά αποτελέσματα. Η Ινδονησία για παράδειγμα και άλλες χώρες ε, οι οποίες ε, ήταν παλαιότερα αλλά δεν είναι πλέον ε, χώρες προέλευσης παρανοής μετανάστευσης. Ε, τι κάνατε για να είσαστε τόσο αποτελεσματικοί στη μείωση αυτών των ροών. Ευχαριστώ. Ωραία. Αυτό ήταν ο πρώτος γύρος ερωτήσεων. Παρακαλώ πολύ. Um, thank you. Thank you very much for... Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις, λέει ο κύριος Άντριους. Από τον... Ε, πρώτη ερώτηση ήταν από τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας. σχέσεις Αυστραλίας με το Ηνωμένο Βασίλειο και με την Ευρώπη. Θα ήταν σωστό να πούμε ότι η Αυστραλία επιδιώκει ένα ελεύθερο εμπόριο βασισμένο σε κανόνες με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή ομάδα χωρών που υποστηρίζει το ίδιο σχέδιο. Αυτό δεν έχει σχέση με το αν θα λάβει χώρα το Brexit ή όχι η προσέγγιση μας δεν αλλάζει. Είμαστε υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και με την ΕΒ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ως συνολικό, συνολικές εμπορικές ροές, το είπα και προηγουμένως, ακόμα και χωρίς το Ηνωμένο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ πιο ισχυρός εμπορικός εταίρος. Δεν υπάρχει συναισθηματισμός ή μάλλον συναισθηματισμός σε θέματα εμπορίου είναι πολύ λίγος. Παίζει πολύ μικρό ρόλο. Εμείς ε, θέλουμε να ενισχύσουμε τις εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πράγματα που θα πρέπει να δουλευτούν όπως σε οποιαδήποτε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Για παράδειγμα ζητήματα που έχουν σχέση με τη γεωργία και τα γεωργικά προϊόντα. Απ' την άλλη μεριά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια θέματα σε σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία, με τις δημόσιες προμήθειες στην Αυστραλία κλπ. Οπότε για μας είναι προτεραιότητα όσο είναι προτεραιότητα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να συνεχίσουμε. Αν επανέλθουμε στη διαπραγματεύση το, το συντομότερο, αυτό θα είναι το καλύτερο. Εμείς ακολουθούμε μια προσέγγιση διεθνή σε ό,τι αφορά το ελεύθερο εμπόριο. Έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά κατανοούμε ταυτόχρονα και τις προκλήσεις. Τώρα, έγιναν ε, ερωτήσεις και για την Κίνα. Για μας η Κίνα είναι και τεράστια ευκαιρία, την οποία έχουμε εκμεταλλευτεί εδώ και αρκετό καιρό, αλλά και πρόκληση. Οι ευκαιρίες έχουν σχέση με την ισχυρή ανάπτυξη της κινέζικης οικονομίας και παρόλο ότι έχει πέσει ο ρυθμός ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια εξακολουθεί να αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από τον υπόλοιπο κόσμο, εξυγχρονίζεται πολύ γρήγορα με ισχυρούς ρυθμούς και θα γίνει ακόμα πιο ισχυρός παίκτη στην παγκόσμια οικονομία. Από την άλλη μεριά δεν είναι μόνο η Κίνα. ο εξυγχρονισμός και η ανάπτυξη λαμβάνουν χώρα σε πολλές άλλες χώρες ε, του ειρηνικού και πολύ συχνά ξεχνάμε και την Ινδία που έχει τεράστιο πληθυσμό και αναπτύσσεται όχι τόσο γρήγορα όσο η Κίνα αλλά εξακολουθεί να έχει πολύ ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αυτό είναι σημαντικό για μας και για όλο τον κόσμο. Σε ό,τι μας αφορά, εμείς επιδιώκουμε έναν ε, ε, εμπόριο, διεθνές εμπόριο βασισμένο σε κανόνες. Κάθε χώρα θα έχει ένα στάτους το οποίο θα προβλέψει συγκεκριμένους κανόνες δικαιώματα και υποχρεώσεις. Είναι πολύ σημαντική η κάθετη ολοκλήρωση σε τομείς όπως η γεωργία, η συνεργασία στον τεχνολογικό τομέα, ε, τεχνολογία 5G, πέμπτης γενιάς, ε, κινητής τηλεφωνίας, ε, επενδύσεις της Κίνας στην Αυστραλία. Θέλουμε όμως όλα αυτά να γίνονται με κανόνες. Η προσέγγιση μας ε, είναι να υποφεληθούμε από τις οικονομικές ευκαιρίες, αλλά να είμαστε και ρεαλιστές σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις. Καθώς επίσης και σε σχέση με τις στρατηγικές πτυχές των σχέσεων αυτών. Ε, όλα τα κράτη της περιοχής, ε, από την Ινδία μέχρι τον Ειρηνικό, έχουν περίπου την ίδια στάση σε ό,τι αφορά την Κίνα. Εμείς ε, είμαστε πιο παρόντες και έχουμε εντείνει τη σχέση μας με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και του Νοτιοανατολικού, συγγνώμη, Ειρηνικού. Και αυτό μας δίνει περισσότερη ισχύ. Τώρα, η καταπολέμηση τρομοκρατίας ε, είναι στοιχιώνει μάλλον της ε, πολιτικής ασφαλείας των κρατών μας. Στην Νοτιοανατολική Ασία φοβόμαστε ιδιαίτερα την επιστροφή ε, ακραίων στοιχείων από την Μέση Ανατολή. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε βέλτιστες σχέσεις με τις κυβερνήσεις της ε, περιφερειάς μας. Ε, και συνεργαζόμαστε όχι μόνο σε θέματα αντιτρομοκρατικά, αλλά και σε ζητήματα που άπτονται των μεταναστεύσεων. Η μετανάστευση αυτή τη στιγμή γίνεται τάξη και αυτό επειδή έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Ινδονησία και τη Μαλαισία συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους σε θέματα μετανάστευσης και συνεργαζόμαστε πολύ θετικά. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, είμαστε πράγματι ένας λαός ε, που προέκυψε από τη μετανάστευση. Το 1 τρίτο του πληθυσμού μας μιλάει στο σπίτι του μια, χώρα, μια γλώσσα που δεν είναι απαραίτητα τα αγγλικά. Οπότε γνωρίζουμε τι είναι η μετανάστευση. Παρ' όλα αυτά, η μεταναστευτική μας πολιτική θα πρέπει να οδηγεί σε μια τακτική μετανάστευση με κανόνες περίπου 160 έως 200.000 ατόμους, ε, ανθρώπους δεχόμαστε ετησίως ως επίσημη μετανάστευση. Και σε οποιοδήποτε, οποιαδήποτε χρονιά έχουμε πάνω από 2 εκατομμύρια προσωρινούς μετανάστες, τουρίστες, ε, φοιτητές, νεοζηλανδοί και μετανάστες με συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα που έρχονται να δουλέψουν στη χώρα μας ε, επί τη βάση προσωρινών προγραμμάτων εργασίας τετραετών ε, και που μπορούν μετά να γίνουν και μόνιμοι κάτοικοι υπό συνθήκες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ε, να πολιτογραφηθούν και Αυστραλοί. Οπότε προσπαθούμε να η μετανάστευση να γίνεται με ένα τακτοποιημένο τρόπο, με κανόνες για συγκεκριμένους τομείς, συγκεκριμένες, συγκεκριμένα προφίλ κλπ. Για τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ασίας. Ε, λάβαμε γνώση τη συμφωνία με την Ιαπωνία. Νομίζω την ε, ψηφίστηκε πολύ πρόσφατα και είμαστε σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να ε, διαπραγματευτούμε ένα πρόγραμμα συνδεσιμότητας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση. Thank you, Kevin Andrews. Ευχαριστούμε, Kevin Andrews. Επόμενος γύρος ερωτήσεων και ξεκινάμε με τον Μιχαήλ Γκάλερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ και καλωσορίσατε και από πλευράς μου η Κινέζικη πριν στην ε, περιοχή αναφέρθηκε ήδη και η ερώτησή μου αφορά ένα ζήτημα που μας αφορά θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία που έχουμε θα λήξει συχνά εμείς έχουμε δραστηριοποιηθεί ε, στην περιοχή, και στην περιοχή όπως και στην περιοχή ΣΥΠΗ. Οι Κινέζοι βάσει ισχυρισμών τους και δραστηριοτήτων τους ε, θεωρείται ότι μπορεί να αναβαθμιστεί η συνεργασία μας στα νησιά αυτά, σε αυτή την περιοχή. Εγώ στο νου έχω κάποια συμπληρωματικότητα, δεν είμαι αφελής. Ε, είναι η δική σας γειτονία, δεν είναι η δική, η δική μας. Εσείς δηλαδή ε, ασκείτε καθημερινή πολιτική στην περιοχή αυτή. Αλλά επειδή τα δικά μας δημοσιονομικά πλαίσια είναι περιορισμένα και έχουμε κάποιες δεσμεύσεις εκεί επίσης, μήπως εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζοντας αυτή την πολιτική στην περιοχή του Ειρηνικού θα πρέπει να συντονιστούμε περισσότερο μαζί σας μήπως ώστε να αλληλοσυμπληρωνόμαστε επειδή έχουμε παρόμοια νοοτροπία, ε, παρόμοιες γενικές κατευθύνσεις. Οπότε μαζί να αντιμετωπίσουμε και τις αρνητικές κινέζικες δραστηριότητες, όχι όλες τις δραστηριότητες, σε καμία περίπτωση το εμπόριο είναι μια χαρά, αλλά τον τρόπο με τον οποίο η Κίνα επιθυμεί να κυριαρχήσει ε, σε ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι σίγουρα δύσκολο για σας, περισσότερο από ότι για εμάς. Αν λοιπόν αναβαθμίζαμε τι δραστηριότητε μας σε αυτόν τον τομέα, μήπω αυτό θα ήταν μια καλή ιδέα για να ε, ασκούμε καλύτερη πολιτική ε, καθημερινά σε, και όχι κατά διαστήματα εδώ. Ευχαριστούμε Μιχαήλ, η κυρία Μοζό και είναι πρόεδρος της Υποεπιτροπής ε, Ασφαλείας και Άμυνας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και από δική μου πλευρά θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τους προσκεκλημένους μα από την Αυστραλία. Πολλοί είμαστε εμείς που θέλουμε να σας θέσουμε ερωτήσεις για τη σχέση σα με την Κίνα. Ποια είναι η άποψή σα για τις κινεζικέ πρωτοβουλίε στο, στο πλαίσιο αυτού που εμείς αποκαλούμε δρόμος του μεταξιού. Οι πρωτοβουλίε αυτές μπορεί να έχουν αντίκτυπο συγκεκριμένο σε στην, στην Ασία. Ποια θα ήταν η γνώμη σας για μια πιο στενή εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας, έτσι ώστε οι Ασιάτες εταίροι μας να έχουν και άλλες επιλογές και να μην ε, υποχρεούνται να μπαίνουν σε ένα μονοπωλιακό διάλογο με την Κίνα. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το διάστημα στο οποίο δραστηριοποιούνται τα κράτη, αλλά δραστηριοποιούνται και εμπορικές επιχειρήσεις και ε, υπάρχει και στρατιωτική διάσταση όλο και περισσότερο. Η Αυστραλία έχει ε, πολύ μακροχρόνιες σχέσεις με την NASA αλλά και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, ε, την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία για την επιτήρηση του διαστήματος. Η Αυστραλία είναι έτοιμη να προχωρήσει ε, με την συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το νέο σύνορο που αποτελεί το διάστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Μπομφρίσκου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε θέλω να πω στην Αυστραλιανή αντιπροσωπεία στα Ιταλικά γιατί έχετε και πολλούς ε, Ιταλικής καταγωγής Αυστραλούς υπηκόους. Αυτό μου επιτρέπει να υπενθυμίσω ότι το αυστραλιανό μοντέλο για τη μετανάστευση είναι πιθανότατα το καλύτερο παγκοσμίω. Δίνει τη δυνατότητα ελέγχου και τακτικής ε, ανάπτυξης οποιασδήποτε μεταναστευτικής πολιτικής. Η ιστορία μας υπενθυμίζει, η δική μας ιστορία μας υποστηρίζει πώς εμείς ε, είχαμε, αμυνθήκαμε από κοινού και είχαμε και την Διατλαντική Συμμαχία της οποίας όλοι είμαστε μέλη και ενώπιον των δυσκολιών ε, σε θέματα ασφάλειας, όπως υπενθύμησαν και άλλοι συνάδελφοι, όπως και η πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμενας. Η ασφάλεια μπορεί να αποτελέσει το έδαφος μιας νέας ανανεωμένης συμμαχίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας. Ο ειρηνικός όλο και περισσότερο αποτελεί αντικείμενο ανησυχία για εμάς. Η ερώτησή μου λοιπόν αφορά ακριβώς αυτό. Ο άκρατος εξοπλισμός της Κίνας και αυτή η επίδειξη ε, πολεμικού υλικού στη σημερινή παρέλαση από την Κίνα σας ανησυχεί και εσάς όπως και εμάς. Το λαό, στους λαούς γενικά και τις ε, κυβερνήσεις της περιοχής και πέραν της άποψης που έχετε σχηματίσει εσείς, έχετε πρόθεση να αναπτύξετε περισσότερο το θέμα της ασφάλειας και της άμυνας, πάντα ακολουθώντα μια λογική ε, διατλαντική συμμαχία, σίγουρα, αλλά και ενδεχομένω με... λαμβάνοντα περισσότερο υπόψη και τις στρατηγικές γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. τελευταίοι δύο στον κατάλογό μου και μετά κλείνουμε είναι ο κύριος Μπένιον και ο κύριος Μαριάννη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν μιλώ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόνο εδώ, αλλά και ως Ευρωπαίος αγρότης. Ως προς τις εμπορικές συμφωνίες, ξέρω από τους συναδέλφους μου στον αγροδιατροφικό και γεωργικό τομέα ότι εκεί επικρατούν πάρα πολλές ανησυχίες. Μεγάλος προβληματισμός ότι μπορεί οι Αυστραλιανοί να πολλούν φθηνότερα ε, ήδη είναι πολύ δύσκολο το περιβάλλον για ένα γεωργό και ένα αγρότη να καταφέρει να σταθεί εμπορικά και να πουλήσει τα προϊόντα του. Γενικά είναι διάσπαρτος ο φόβος. Και αυτό οξύνεται και με τα θέματα του Brexit ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι σίγουρα υπάρχει ένα στοιχείο διασπαστικό εντός της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, η οποία προτείνει μηδέν δασμούς για το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Μηδέν εισερχόμενους δασμούς παγκοσμίω. Είναι μια ομάδα βουλευτών που ουσιαστικά θέλουν να παρακολύσουν την παγκόσμια τάξη πραγμάτων στο πλαίσιο του ΠΟΕ και συμφωνούν με την ατζέντα του Ντόναλτ Τραμπ. Ε, το αντεπιχείρημα όμως είναι ότι η Αυστραλία και η Νέα ε, Ζηλανδία από κοινού ουσιαστικά δεν μπορούν να πλημμυρίσουν τις αγορές μας με πάθυνα προϊόντα, ακόμα και αν θα το ήθελαν, διότι συγκεντρώνονται και επικεντρώνονται ούτως ή άλλως στις ασιατικές αγορές πρώτον και δεύτερον ε, διότι η παραγωγική τους ικανότητα είναι πολύ μικρή συγκριτικά με το παραγωγικό δυναμικό της Ευρώπης. Ήθελα τη δική σας άποψη για αυτά, δηλαδή σε ποιο βαθμό Μία εμπορική συμφωνία θα λειτουργούσε διασπαστικά στη δική μας ε, βιομηχανία, ε, λαμβάνοντας αυτά τα θέματα υπόψη. Είχα και ένα δεύτερο ερώτημα για την Κίνα, αλλά άκουσα όλους να θέτουν ερωτήματα για την Κίνα ούτως ή άλλως. Δύο είναι οι γεωπολιτικές πτυχές με την Κίνα που μας ανησυχούν και μας προβληματίζουν. Η κατάσταση στη θάλασσα της Νότιας Κίνας, όπου έχουν ε, ε, διεκδικήσεις ε, από τις όμορες και γειτονικές τους χώρες σε σχέση με το ζωτικό τους χώρο. Αυτό είναι υπερβολικό, είναι πολύ μακριά από εσά για να σας ανησυχήσει. Ποια είναι η στάση σας για το θέμα της θάλασσας της Νότιας Κίνας και το θέμα του δρόμου του μεταξιού. Η Κίνα χρησιμοποιεί την οικονομική της δύναμη απευθυνόμενη στις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες οφείλουν στην Κίνα και αξιοποιεί αυτά τα χρέη για να επιτύχει τις πολιτικές της επιδιώξεις. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό, στηρίζω τους προλαλήσαντες. Ίσως θα έπρεπε να ευθυγραμμιστούμε με πιο στρατηγικά έξυπνο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Ο κύριος Μαριάννη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συμφωνία που μας προτείνεται έχει ως στόχο να θεσπίσει μια ανισχυμένη εταιρική σχέση και να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να ενθαρρύνει τη συνεργασία σε πλειάδα ε, κοινών ενδιαφέρων και επιδιώξεων. Θέλω να σταθώ σε δύο σημεία και θέλω να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Όπως λέει η συμφωνία θα ήταν επιθυμητό και ευκταίο εμπιστευτικές πληροφορίες να ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Όμως οι υπηρεσίες ασφαλείας κάθε κράτους έχουν έχουν την αρμοδιότητα για να διευθετήσουν αυτό το πρόβλημα και από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει αντιτρομοκρατική υπηρεσία ευρωπαϊκή. Άρα αυτή η συμφωνία για άλλη μια φορά δεν χρησιμεύει παρά μόνο στο να υπεξαιρέσει την εθνική κυριαρχία των κρατών και ε, σε αυτή τη, το συγκεκριμένο παράδειγμα της ανταλλαγής πληροφοριών πώς θα λειτουργήσει τάχα μου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία αφού, ευρωπαϊκές, αφού εθνικές κρατικές υπηρεσίες ανταλλάσσουν αυτές τις ε, πληροφορίες και δεν έχει Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Αντιτρομοκρατική. Από εκεί και πέρα, ε, για τη μετανάστευση θα ήθελα να γνωρίσω εάν προβλέπετε συνεργασία ανταλλαγή πληροφοριών με την υπηρεσία Frontex διότι σε αυτό το επίπεδο πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όντως αρμοδιότητα και καλώς. Και δύο λόγια προσωπικά θέλω να πω, γιατί είμαι πρώην ε, μέλος του Γαλλικού Κοινοβουλίου που έχω εκλεγεί από τους Γάλλους ομογενείς του εξωτερικού. Ε, για γι' αυτό έχω επισκεφθεί τη χώρα σας ε, πάρα πολλές φορές ε, τουλάχιστον 30 και δεν θέλω να ξεχνάτε τις θυσίες των Γάλλων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να ε, απαντήσω μαζί κάποιες ερωτήσεις. Πολλές αφορούσαν την Κίνα και χωρίς να θέλω να επαναλάβω αυτά που είπα προηγουμένως. Πιστεύω είναι σημαντικό για κάθε χώρα που θέλει να συνεχίσει να έχει καλές σχέσεις με την Κίνα να επισημάνει στην Κίνα ότι δεν συμφέρει μόνο εμάς αλλά και την Κίνα να μπορούμε να, να την κατανοούμε και να ακολουθούν ένα σύστημα ε, συμφωνημένο παγκόσμιο κανόνων. Αυτό θέλουμε εμείς να κάνουμε την Κίνα και θέλουμε και εσείς να το επισημαίνετε στην Κίνα. Όπου έχουμε περιπτώσεις, ε, πώς να το πω, όπου φλερτάρει κάποιος κάποια άλλη προσέγγιση, αυτό θα πρέπει να ακολουθούμε. Ε, αυτό που μας λέει η ιστορία είναι ότι αν δεν υπάρχει κάποια τάξη βασισμένη σε κανόνες ε, μπορεί να υπάρχουν απρόβλεπτες συνέπειες οι οποίες δεν είναι μονομερείς ε, επηρεάζουν όλα τα μέρη με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Η επιχειρηματολογία μας λοιπόν μπροστά στην Κίνα είναι ότι συμφέρει την ίδια την Κίνα όπως συμφέρει και εμάς και τον κόσμο ολόκληρο να συμφωνήσουμε, να συμφωνούμε για μια διεθνή προσέγγιση αυτό αφορά ζητήματα όπως την ε, Νότια Θάλασσα της Κίνας, ε, ζητήματα ε, οικονομικού, οικονομίας εμπορίου και άλλους τομείς. Ήθελα επίσης να πω ότι η Κίνα δεν είναι απλά μια γείτονα χώρα της Αυστραλίας. Αφορά οι σχέσεις μας με την Κίνα όλο τον κόσμο. Και αυτό θα εντείνεται στο μέλλον, πιστεύω. Η Ευρώπη μπορεί να απέχει λίγο παραπάνω από την Κίνα όσον αφορά τι άμεσε δραστηριότητες από την Αυστραλία. Παρ' όλα αυτά, ό,τι συμβαίνει στις σχέσεις Αυστραλίας και Κίνας και άλλων χωρών και Κίνας θα επηρεάσει όλους μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό είναι σημαντικό, επαναλαμβάνω, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ούτω ώστε να μπορούμε να επιλύουμε ειρηνικά οποιαδήποτε προβλήματα ενδεχομένως προκύψουν σε θέματα νησιών ή επίσημων δομών, όπως και να το ονομάσουμε στη Νότια Θάλασσα της Κίνας. Διότι ξέρετε, το παγκοσμίο εμπόριο κυκλοφορεί πάνω σε διάφορε υδάτινε οδού και κάτι, ε, προβλήματα εκεί θα επηρεάσουν την ευημερία για όλου, και για την Ευρώπη και για την Αυστραλία και για την Κίνα. Όπω είπα νωρίτερα, η Κίνα αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για εμά, αλλά δημιουργεί και διάφορες ε, προκλήσεις και πρέπει να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε όλα αυτά ούτως ώστε να συνεχιστούν οι συνομιλίες με την Κίνα για τα θέματα που συμφέρουν όλους μας και εμάς και την Ευρώπη. Ακούσαμε κάποιες άλλες ερωτήσεις για τη μετανάστευση και την προσέγγισή μας της μετανάστευσης. Εμεί είμαστε ικανοποιημένοι ε, από αυτή την προσέγγιση. Μέσω τη πρεσβεία μα εδώ στι ε, Βρυξέλλε και των άλλων πρεσβειών μα, θέλουμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για την προσέγγιση αυτή. Κάθε χώρα είναι μοναδική από πολλέ απόψει. Ε, εμείς εκεί που βρισκόμαστε ως νήσος ουσιαστικά τη μετανάστευση την αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Δεν υπάρχει λοιπόν μια λύση που να βολεύει όλους. Ούτε θα ήθελα να προτείνω κάτι τέτοιο ή να πω ότι η δική μας λύση είναι μοναδική και ότι όλοι πρέπει να κάνουν το ίδιο. Αλλά σίγουρα μια διαδικασία βασισμένη σε κανόνες είναι σημαντική και για μια χώρα όπως η Αυστραλία που εξαρτάται ε, εδώ και δεκαετίες από τη μεταναστεύση και θα συνεχίσει και στο μέλλον. Χωρίς μια τέτοια διαδικασία βάση κανόνων υπάρχει ε, το ενδεχόμενο απρόβλεπτων συνεπειών για τη χώρα μας και ουσιαστικά και για άλλες. Όσον αφορά τη γεωργία και τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών, ήθελα να πω ότι ως γιος αγρότη, παντρεμένο με κόρη αγρότη, εκτιμώ τις ανησυχίε των αγροτών όπου και αν ζουν στον κόσμο σε σχέση με τη γεωργία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συνεννόηση αμοιβαία εποφελή. Για τη δική μας χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν οι προοπτικές παγκοσμίω με την αύξηση του πληθυσμού και την αύξηση της μεσαίας τάξης είναι ότι θα αυξηθεί η ζήτηση γεωργικών προϊόντων αντί να μειωθεί. Αν καταλήξουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα υποφελεί τους ε, Ευρωπαίους και τους Αυστραλούς γεωργούς, αυτό θα επιδιώξουμε και εμείς. Εμείς θέλουμε μια δίκαιη διαδικασία που θα ωφελεί εμάς, αλλά όπως καταλαβαίνουμε πρέπει να υποφελεί και την Ευρώπη με αυτό το πνεύμα θα μπούμε σε οποιασδήποτε διαπραγματεύσει ελεύθερων συναλλαγών. Μη θυμάστε ότι τα γεωργικά προϊόντα απάντα αποτελούν σημαντικό διακύβευμα και στην Αυστραλία και στην Ευρώπη. Μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών θα αφορά πολλά περισσότερα από απλά ε, τα γεωργικά προϊόντα. Σε ένα κόσμο γεμάτο υπηρεσίε ε, ε, ενέχει διάφορε άλλε ευκαιρίε επίση σε θέματα αυτό προβλέπουμε και μια συμφωνία ελευθερών συναλλαγών στο μέλλον. Ε, τέθηκε το ερώτημα της Ευρωπαϊκής, της, των δραστηριοτήτων Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ειρηνικό και στον Νότιο Ειρηνικό ειδικότερα. Εμεί καλωσορίζουμε οποιαδήποτε συνεργασία για μια καλύτερη παρουσία, να βοηθήσουμε να ε, υπάρχει τέτοια δραστηριότητα ε, ειδικότερα στα νησιά του Νοτιού Ειρηνικού να δούμε τι γίνεται με τις παγίδες που στην η Κίνα εκεί πέρα σε αυτά τα νησιωτικά κράτη. Ξέρετε, υπόσχονται ένα νοσοκομείο, ένα δρόμο σε ένα μικρό κράτο, νησιωτικό κράτο εκεί και αυτοί το βρίσκουν ελκυστικό, χωρί να αντιλαμβάνονται ακριβώ ποιε είναι οι απότερε συνέπειε. Όσον αφορά την πρωτοβουλία Μια Ζώνη, ένα δρόμο, είναι σημαντική αλλά πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ τη ρητορική δημοσίων σχέσεων και τη πραγματική απόδοση, δωρεπιδόσεων μια τέτοια πρωτοβουλία. Έχουν ε, κάνει πολλά σε θέματα δημοσίων σχέσεων, αλλά σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι οι αποδόσει είναι τόσο καταπληκτικέ ή ότι αντιστοιχούν στη ρητορική που ακούμε. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ, ε, υπερασπιζόμενοι τα δικά μα και τα δικά σα συμφέροντα. Το θέμα είναι και πάλι να καταλάβουμε καλά, να έχουμε κανόνε ε, του οποίου έχουμε συνεννοηθεί, του οποίου κατανοούμε, οι οποίοι είναι καθαροί, ώστε να ευημερούν όλε οι χώρε και η Κίνα. Και μετά, άλλη μια ερώτηση. Νομίζω ότι κάλυψα τι περισσότερε. Ακούσαμε μια ερώτηση για την ανταλλαγή ε, απορρίτων πληροφοριών. Έχουμε πράγματι τακτικές ε, διαβουλεύσεις για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας με την Ευρώπη και με τους μεγαλύτερους ε, φορείς ασφαλείας στην Ευρώπη, ασφαλείας στην Ευρώπη με γνώμονα την αντιμετώπιση των κοινών απειλών. Έχουμε μια διμερή συμφωνία που προβλέπει ανταλλαγή κάποιων ε, διαβαθμισμένων πληροφοριών και η συμφωνία αυτή λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. Φυσικά οποιαδήποτε ευκαιρία βελτίωσης ε, μιας τέτοιας συμφωνίας ε, και των ε, συναφών συμφωνιών μας βρίσκει σύμφωνο. Εμείς πάντα είμαστε διατεθειμένοι να συνομιλήσουμε μαζί σας για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τέτοιες συμφωνίες. Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι ένα μεγάλο ζήτημα παγκοσμίω και θα εξακολουθήσει να είναι μέσα στα επόμενα χρόνια και τις δεκαετίες. Ευχαριστώ. Κέβιν Άντριου, σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις που δώσατε. Θα ευχαριστώ ευχαριστήσουμε και τους ε, συναδέλφους σας από την Αυστραλία που ήρθαν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Τρεις ε, τελικές παρατηρήσεις από πλευράς μου. Παρακαλούμε πρώτον, συνεχίστε να απολαμβάνετε την πολυμορφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Έχουμε 751 ε, συναδέλφους από 28 χώρες, 7 πολιτικές ομάδες και 24 διαφορετικές γλώσσες. Πήρατε μια γεύση σήμερα ε, για την πολυμορφία των απόψεων ε, και των ε, διαφορετικών καταγωγών που έχουν εδώ οι συνάδελφοι. Το δεύτερο, οι συνάδελφοι φυσικά έχουν και επαφές με συναδέλφους από άλλες αγγλόφωνες χώρες. Εάν βρεθείτε σε Βρετανούς συναδέλφους που υποστηρίζουν το Brexit, να είστε πολύ προσεκτικοί. και καταρρύψτε τα επιχειρήματά τους, γιατί δεν βασίζονται 100% σε γεγονότα, οι οι ε, Βρετανοί μα συναδέλφοι μερικές φορές ε, ε, λένε πράγματα αρκετά ανακριβή όσον αφορά το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να σε ευχηθούμε καλή τύχη για το επόμενο μάτς του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράγκμπι. Θα παίξει η Αυστραλία με την Ουρουάη και είναι σημαντικό το μάτς αυτό γιατί χάσατε για λίγο με την... από την Ουαλία αυτό το Σαββατοκυριακό. Οπότε καλή τύχη. Ελπίζουμε να σας δούμε στους ημιτελικούς ή και καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you. We are the same organization. Yes. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συνεχίσουμε με την πρωινή μας συνεδρία. Ερχόμαστε στο σημείο 6. Να καλωσορίσουμε θερμά την κυρία Τζόις Μεσούγια. Δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομά σας. Πολύ σωστά το προφέρετε. Καλωσορίσατε, κυρία Τζόις Μεσούγια από τα Ηνωμένα Έθνη είναι βοηθός γενική γραμματική ε, και εκτελεστική διευθύντρια του περιβαλλοντικού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών. Η παρουσία της κυρίας Μεσούγια στην σημερινή μας συνεδρίαση έρχεται σε, ένα σε μια πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία μετά την ε, τελευταία σύνοδο στον για το κλίμα που ολοκλήρωσε τις εργασίες της χθες. 30 Σεπτεμβρίου. Παρακολουθήσαμε όλοι στενά τις συζητήσεις στη Νέα Υόρκη. Η κλιματική δράση αποτελεί μέρος των δεσμεύσεων του Γενικού Γραμματέα Γκουτιέρες για την προώθηση μιας παγκόσμιας πολιτικής για την προστασία του κλίματος. Όλα αυτά τονίζουν τη σημασία της πολυμέρειας, της πολυμερούς ανταπόκρισης στα προβλήματα και έτσι η, ε, θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το πρόβλημα. Πώς ερμηνεύει ο ΙΕ την κατάληξη της συνόδου αυτή για το κλίμα, ποια θα είναι η συνέχεια που θα δοθεί, ποιες είναι οι οι προσδοκίες σας για το μέλλον αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να υπάρξει συνένεση και μεγαλύτερη συμμετοχή για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και για τη συνέχιση του διαλόγου για τις διάφορες περιφέρειες οι οποίες κινδυνεύουν περισσότερα από την υποβάθμιση ε, της κατάστασης σε σχέση με το κλίμα, η Λατινική Αμερική, Ασία η Αφρικανική υπήρξη μεταξύ άλλων. Θα ήθελα να σα δώσω το λόγο και μετά θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους. Καλώ ορίσατε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μακάλιστερ. Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ μαζί σας για να σας μιλήσω. Εκ μέρους του Οργανισμού Εθνών σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θερμά, για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε. Θα εστιάσω σε τρεις πτυχές, σύμφωνα με τις οδηγίες που μου έδωσε ο κ. Μακάλιστερ. Πρώτον, θα σας μιλήσω για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής για το κλίμα, της διάσκεψης κορυφής για το κλίμα. Δεύτερον, τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Και τρίτον, θα απαντήσω σε δικές σας ερωτήσεις. Καταρχήν σε ό,τι αφορά την ε, διάσκεψη κορυφή του ΕΕ για το κλίμα. Όπω είπε και ο Γενικό Γραμματέα κ. Γκουτέρε, η διάσκεψη αυτή είχε στόχο στο να καταλήξουμε σε φιλόδοξα σχέδια και δράσει από πλευρά των κυβερνήσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και από την πλευρά ε, του ιδιωτικού τομέα, με κυβερνητικών οργανώσεων και ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Είδαμε ένα πολύ ισχυρό δυναμισμό και προσήλωση σε αυτό το έργο, καθώς επίσης και αρκετή ανυπομονησία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια πολύ σημαντική παρουσία υπέρ της πολυμέρειας, της πολυμερούς ε, δράσης και η, και η όλη διάσκεψη κατέδειξε την ισχύ της πολυμέρειας διότι έφερε στο ίδιο τραπέζι όλους τους παίκτες για να συζητήσουν την πιο σημαντική ενδεχομένως πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, την κλιματική αλλαγή. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα λοιπόν, 65 χώρες και τμήματα χωρών όπως η Καλιφόρνια ανέλαβαν την ευθύνη να μειώσουν μέχρι το 2050 στο 0 τις εκπομπές τους και 17 χώρες ανακοίνωσαν ότι ή θα ενισχύσουν τα εθνικά τους προγράμματα μέχρι 2020 ή θα ξεκινήσουν τη διαδικασία να κάνουν κάτι τέτοιο. Και συνεργαζόμαστε πολύ στενά με αυτές τις τελευταίες έτσι ώστε να επιταχύνουν. Πάνω από 100 επιχειρηματίες επίσης ε, ανακοίνωσαν συγκεκριμένες δράσεις σύμφωνες με τους στόχους του Παρισιού και προκειμένου να περάσουμε γρήγορα στην πράσινη οικονομία. Ε, μεταξύ αυτών ε, ε, και ε, επιχειρηματίες που διαθέτουν ποσά πάνω των 2, των 3 εκατομμυρίων δολαρίων. 87 εταιρείε με κεφαλαίο, συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων ε, ανακοίνωσαν ότι θα μειώσουν τις εκπομπές τους μέχρι το 2050. 130 τράπεζες, το 1 τρίτο δηλαδή του συνολικού παγκόσμιου τραπεζικού τομέα, υπέγραψαν τη συμφωνία ε, προκειμένου οι επιχειρήσεις τους να ευθυγραμμιστούν με τους στόχους του Παρισιού. Οπότε τεράστιος ο αριθμός ε, των δεσμεύσεων που ελήφθησαν και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνείς παίκτες και ενδιαφερόμενους φορείς. Τώρα, τι σκοπεύουμε να κάνουμε στο μέλλον. Αμέσω μετά την επισκεψή μου εδώ στι Βρυξέλλες ε, θα ξεκινήσουμε τα προγράμματα δράση που θα ακολουθήσουν έτσι ώστε αυτέ οι δεσμεύσει να γίνουν πράξη, να υλοποιηθούν. Σε επίπεδο ΟΗΕ αυτό θα γίνει σε στενή συνεργασία με, την, με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα και με τα γραφεία των βοηθών Γενικών Γραμματέων. Σε εθνικό επίπεδο, μέσω των υπηρεσιών του ΟΗΕ, θα δούμε πώς ο ΙΕ ως σύνολο, συνολικά, ως οργανισμός μπορεί να στηρίξει τις χώρες έτσι ώστε να ελοπίσουν τις δράσεις τους. Τις, ε, ε, για παράδειγμα, ο Γενικός Γραμματέας μας ζήτησε να παρακολουθήσουμε το πώς η φύση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα τα δάση λάβαμε ένα πολιτικό μήνυμα, λάβαμε ένα πολιτικό ε, ε, στίγμα στη Νέα Υόρκη και μαζί με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε τον ιδιωτικό τομέα, τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και άλλε διεθνεί οργανώσει εκτό του ΟΗΕ προ αυτή την κατεύθυνση. Θα δημιουργήσουμε μια ομάδα φίλων που θα έχει ένα πρόγραμμα δράσης 18 μηνών με πολύ συγκεκριμένα παραδοτέα ε, που θα οδηγήσουν ε, στην ε, χρήση, σε ένα μανιφέστο που θα έχει σχέση με την χρήση της φύσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ο ρόλος των δασών, για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί πόσο ωφέλιμος και κρίσιμος μπορεί να είναι. Θα δώσουμε λοιπόν συνέχεια και θα ενισχύσουμε τα προγραμματά μας για την δάσωση σε διάφορες χώρες του πλανήτη. Θα διοργανώσουμε στις Βρυξέλλες και μία εκδήλωση ε, που η, τις οποίες την οργάνωση θα αναλάβει το γραφείο μας εδώ και η Βερόνικα. Εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς θα προσκληθούν ε, να συμμετάσχουν. Ε, και εγώ είμαι στη διάθεσή σας, αλλά και η ομάδα μου οποιαδήποτε στιγμή αφού φύγω εγώ. Κύριε Μακάλιστερ, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μεσούγια, για τις παρατηρήσεις σας, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα ξεκινήσουμε με τις πολιτικές ομάδες με τη σειρά τους. Από τους σοσιαλιστές καταρχήν ο κύριος Λόπες. Presidente, yo Ευχαριστώ πολύ. Δύο σχόλια έχω να κάνω. Και μια ερωτσούλα. Καταρχήν, είχα την τύχη να είμαι μέλος της ε, Επιτροπής του Κοινοβουλίου στην ε, Νέα Υόρκη. Εγώ εκ μέρους της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, και παρακολούθησα και τις δύο διασκέψεις και της βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής διάσκεψης. Εργαστήκαμε πολύ καλά και πολύ στενά με διάφορους επιτρόπους που ήταν επίσης παρόντες ε, και με τον πρέσβη μας στις ΗΠΑ. Οπότε η δική μας παρουσία και συμμετοχή ήταν δυναμική, ήταν συνεχής. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Ως ε, καρπός αυτής της συμμετοχής πέραν το ότι αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις, ε, να τηρήσουμε τους στόχους του Παρισιού, να κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια τα επόμενα δέκα χρόνια για να ε, αποκτήσουμε μέχρι το 2050 μια οικονομία που θα έχει μηδενική συνεισφορά άνθρακα. Θέλω, πέραν αυτών λέω, να κάνω κάποιες σκέψεις σε ό,τι αφορά ε, την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνής μας σχέσης. Ποιε είναι αυτές οι σκέψεις. Σε ό,τι φορά καταρχήν το ρόλο των ΗΕ. Είναι πολύ σημαντικό που, το ενωμένο, που ο Οργανισμός έχει αναλάβει μια ηγετική θέση για αυτό το πρόβλημα παρόλο ότι η αποστολή του ΟΗΕ είναι να διατηρεί την ειρήνη. Ε, όμως η κλιματική αλλαγή είναι μια απειλή που εναντίον της ειρήνης και δεν είναι τυχαίο που ένας Ευρωπαίος είναι αυτή τη στιγμή επικεφαλής του ΟΗΕ και ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Δεύτερον, δεύτερη σκέψη. Η πολυμερής προσέγγιση χρειάζεται επιχειρήματα υπέρ της, διότι έχει πληγή βαθιά. Ε, τρίτον, η Ευρώπη ηγείται αυτή του διαλόγου αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ηγείται πολύ λίγων προσπαθειών στον κόσμο. Αυτή, αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα. Τέταρτον, για μας είναι πολύ σημαντικό γιατί η ζωή μας εξαρτάται από αυτό. Όμως γεωπολιτικά έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία η καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής διότι μέσω αυτού μπορούμε να καταργήσουμε την ενεργειακή μας εξάρτηση και δεύτερον, στον τεχνολογικό πόλεμο έχουμε χάσει πολλές μάχες. Από τις 100 μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου, μόνο 8 είναι ευρωπαϊκές. Κίνα και οι και Ηνωμένε Πολιτείε είναι στι πρώτε θέσει. Και μπορούμε μέσω τη δράση μα για το κλίμα να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Τη τεχνολογική υστέρηση. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Λόπε. Πάμε τώρα Ήταν εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι ακούσαμε από το Γενικό Γραμματέα τον κύριο Κουτιέρε τα εξής λόγια, ότι οι χώρε που ήρθαν στα ΟΝΟΙΕ δεν ήρθαν έτοιμε να εκφωνήσουν ομιλίες, έφεραν μαζί τους την πραγματικότητα που βιώνουν. Αυτό δείχνει πόσο ρεαλιστικά αντιμετωπίζει την κατάσταση ο Γενικό Γραμματέα. Όμω, με ομιλίε ήρθαν και ο καθένα ήθελε να παρουσιάσει τη δική του πραγματικότητα. Η κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει μόνο ότι χώρε όπω το Κυριμπάτι, η Μαλτίβε, το Τουβαλού και άλλε ε, τέτοιου είδου χώρε θα εξαφανιστούν από το χάρτη. Είναι και, το, είναι και ένα πρόβλημα στρατηγική ασφάλεια το πρόβλημα τη κλιματική αλλαγή. Η ΙΠΑ είναι από τι χώρε που εκπέμπουν ε, τα περισσότερα αέρια που ευθύνονται για το φαινόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου που οδηγεί στην κλιματική αλλαγή και βρίσκονται σε φάση αρνητισμού. Έχουμε πολύ πικρές πραγματικότητες, μια πολύ πικρή πραγματικότητα και πάρα πολύ ωραία λόγια και εξαιρετικέ ομιλίες. Η Κίνα έχει μια αντιμετώπιση για την ε, στρατηγική με, η οποία η οποία είναι πάρα πολύ αμφισβητούσιμη. Στο ε, ποταμό Βραχμαπούτρα ε, ουσιαστικά παρεμβαίνει η Κίνα και έχουμε την ε, έλευση στερεών υλικών στο Δέλτα, το οποίο ουσιαστικά σε αυτό οφείλεται η ασφάλεια και η υγεία στον Μπαγκλατές. Ουσιαστικά άνθρωποι θα ε, εξαφανιστούν διότι θα προχωρήσει η θάλασσα, θα έχουμε διάβρωση των εδαφών ε, λόγω της αφαλάτωσης και όλων αυτών των δραστηριοτήτων. Και άρα αυτό θα επηρεάσει και την ασφάλεια στην Ινδία, όπου δεκάδες εκατομμύρια μουσουλμάνοι από τον Μπαγκλαντές αναγκαστούν να γίνουν πρόσφυγες και να μπουν στη Βεγγάλη και αλλού, όπου ε, σε παρελθούσες δεκαετίες είχαμε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες, ακριβώς λόγω αυτής της σύγκρουσης. Επομένως δεν σας μιλώ μόνο για τη ρήπανση, για τα προβλήματα αναπνευστικά, για τη μόλυση του περιβάλλοντος, για το, ε, τη θαυμαστή βλάστηση της Αμαζονίας που χάνεται, αλλά μιλώ και για ε, θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Εξαφανίζεται η, τροπική ε, ζώνη, το τροπικό δάσος και στον σημερινό λοιπόν τα εδάφη και οι γέες θα είναι πάρα πολύ ευπαθή. Ουσιαστικά η βλάστηση είναι αυτή η οποία κρατάει το έδαφος και διατηρεί την τροπική ε, ζώνη ε, στο κόσμο περιμετρικά και γι' αυτό έχουμε τα διαφορετικά κλίματα στη ε, ζώνη του καρκίνου και του εγώκερου. Επειδή ακριβώς υπάρχει ισορροπία στη ζώνη στο κέντρο του πλανήτη, στην περίμετρό του, πρέπει να ασχοληθούμε με την πραγματικότητα. Και σας το λέω από τα βάθη της καρδιάς μου. Ε, ε, πια έχουμε αποκτήσει από τις όμορφες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα και όλων των λοιπόν αρμοδίων ε, και έχουμε φτάσει σε απόγνωση από την πολύ άσχημη πραγματικότητα που βιώνουμε. Ευχαριστώ. Για την κούρση, συνάδελφος κ. Βόλας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Οι οικονομικές κυρώσεις είναι ένα αργό βασανιστήριο και οι είναι ένα εργαλείο για να αλλάξει η κυβέρνηση, αλλά ακροτηριάζουν και τις προσπάθειες μείωσης ε, των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Στο Ιράν, ας πούμε, θα μπορούσαν να παράγουν καύσιμο, ε, θα μπορούσαν να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου. Το δικό τους πετρέλαιο θα μπορούσε να περιέχει λιγότερα ε, τέτοια αέρια, να παράγεται λιγότερα τέτοια αέρια από ό,τι αυτό που εισάγουν το Ιράν έχει επιταχύνει τη ε, υδρολογικά έργα για να διασφαλίσει και την διατροφική ασφαλεία λόγω των ε, αμερικανικών κυρώσεων. Αυτό οδήγησε σε σημαντική υποβαθμίση των υπόγειων υδάτων. Ανώ από το 70% των υπόγειων υδάτων του Ιράν έχουν χαθεί ανεπανόρθωτα ε, στην COP21 το 2015 δεσμεύτηκε το Ιράν να μειώσει τις εκπομπές και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 4% ε, εάν δεν ε, ε, επιβάλλονταν κυρώσεις. Επιβλήθηκαν όμως. Μήπως ανησυχείτε αυτές οι κυρώσεις εμποδίζουν μήπως τις χώρες αυτές να προβούν στις αλλαγές που είναι απαραίτητε για την πρόθεση των βιώσιμων κλιματικών πολιτικών. Και πείτε μου αυτό συζητήθηκε στην Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Wallace. Δύο ακόμα. Next is our colleague. Η κυρία Φωνβίζε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ σήμερα από την Σύνοδο Κορυφή για το Κλίμα των Ηνωμένων Εθνών. Εγώ προέρχομαι από την εκλογική περιφέρεια του Λονδίνου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και οι ψηφοφόροι μου ρωτούν το εξή: Τι κάνουμε όσον αφορά την κλιματική δράση. Προφανώ θα θέλαμε Θα θέλαμε όλα τα κράτη-μέλη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να δεσμευτούν για ε, ουδέτερε οικονομίε προ τον άνθρακα μέχρι το 2050. Αλλά η ερώτησή μου είναι, όταν έχουμε εθνικέ κυβερνήσει οι οποίε δεν δεσμεύονται για του στόχου ε, περιορισμού τη κλιματική αλλαγή, Είπατε εσεί ότι υπάρχουν υποεθνικέ ενότητε, οντότητε, όπω περιφέρειε, όπω Καλιφόρνια, που έχουν δεσμευτεί ανεξαρτήτω τη ε, εθνική κυβέρνηση. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, την οποία μπορούμε να ακολουθήσουμε και εμεί αλλού. Ε, περιφέρειες αλλά φυσικά όχι μόνο και ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν διότι ενδεχομένως έχουν ε, ίδια ή και μεγαλύτερη εξουσία και δύναμη να μειώσουν τις εκπομπές τους. Αυτό θα μπορούσαμε να το επιδιώξουμε ως μοντέλο και στην Ευρώπη όπου κάποιες περιφέρειες, κάποιες περιοχές μπορεί να θέλουν να επιταχύνουν, να προχωρήσουν πιο φιλόδοξα από ό,τι άλλες. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστούμε κυρία Φονβίζα.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 είναι ότι οι προσδοκίες ε, ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί του τομέα αυτού από διάφορες γενιές, νέους ε, και από άψη πολιτικής είναι τεράστιες. Επίσης υπάρχουν προσδοκίες να αποτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μοντέλο ως ηγέτης σε επίπεδο πολυμορφίας να καθοδηγεί την παγκόσμια ατζέντα για τα ε, δημόσια αγαθά ε, και να ηγηθεί και της ε, κλιματικής αλλαγής, η οποία δεν έχει γεωγραφικά σύνορα. Από πλευρά μα έχουμε μακροχρόνια συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από του λόγου που βρίσκομαι εδώ είναι να συζητήσω με διάφορε διευθύνσει και ευρωβουλευτέ για να δω τι κάνουμε καλά, τι μπορούμε να αναβαθμίσουμε και να βελτιώσουμε. Αλλά σαφώ παγκοσμίω συμφωνώ μαζί σα οι ευκαιρίες που υπάρχουν μέσω της κλιματικής διπλωματίας είναι τεράστιες ε, να εντάξουμε στον κύριο άξονα των πολιτικών το περιβάλλον και σε παγκόσμιο και σε ε, επίπεδο και σε επίπεδο χωρών. Αναμένω λοιπόν να ανταλλάξουμε ιδέες και να συνεχίσω να έχω την υποστήριξη του Κοινοβουλίου εδώ για να μπορέσετε να μας βοηθήσετε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να κάνουμε κάτι ξεχωριστό και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς του νέου τους νέους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ που θέσατε το θέμα των Κυριμπάτη και την ασφάλεια. Ένα από τα προγράμματα που έχουμε εμεί αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο πρόγραμμα των Ηνωμένων για το περιβάλλον αυτή η διασύνδεση μεταξύ περιβάλλοντος και ασφάλειας. Αν δείτε παγκοσμίω, είτε λόγω ξηρασία, είτε λίγο αποδάσωση ε, ή παρόμοιων προβλημάτων, τα ζητήματα τη ασφάλεια βρίσκονται στο επίκεντρο. Πρέπει να βοηθήσουμε να ενημερώνονται οι αρμόδιοι εξωτερική πολιτική σε ορισμένε ε, χώρε. Ε, και εδώ η υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε σημαντική. η πρόοδο που βλέπουμε σε κάποιε χώρε μα ενθαρρύνει. Έχουμε τα στοιχεία και μπορούμε να τα μοιραστούμε μαζί σα. Για παράδειγμα, η έκθεσή μα για το χάσμα εκπομπών ε, βλέπουμε βάσει αυτή τη έκθεσης ότι σε πολλές μηχανοποιημένε χώρε, όσον αφορά τη ρήπανση σημειώνεται πρόοδο. Παρ' όλα αυτά δεν πάει να αποτελεί πραγματικότητα ότι κάποιε μεταβάσει από μη καθαρέ πηγέ ενέργεια σε καθαρέ πηγέ ενέργεια είναι κάτι χρονοβόρο. Τι κάνουμε εμείς, χρησιμοποιούμε τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας και τις νομοθεσίες μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να επιταχυνθεί αυτή η δράση. Εγώ θα έλεγα από τη Συνόδο Κορυφής για το κλίμα η τεράστια συμμετοχή νέων ανθρώπων δίνει μια διαφορετική διάσταση και διαφορετική ορμή. Πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Για τα μικρά νησιά το παρακολουθούμε. Έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα υπό τον Γενικό Διευθυντή επί το Γενικό Γραμματέα για τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη. Ε, συγγνώμη, για τα μικρά αναπτυσσόμενα κράτη και αυτό, αυτά περιλαμβάνουν πολλά νησιά. Ο Γενικός Γραμματέας είπε ο χρόνος εξαντλείται, η κλιματική αλλαγή είναι ταχύτερη από τις δράσεις μας και δεσμευόμαστε να προωθήσουμε τα πράγματα γνωρίζοντας επίσης ότι ε, τη δράση θα την διαχειριστούμε σε ε, επίπεδο χώρο ουσιαστικά, αλλά και στο δικό μα επίπεδο προσπαθούμε να επιταχύνουμε. Ακούσαμε και μια ερώτηση από ένα μέλο για το κατά πόσο οι κυρώσει στο Ιράν συζητήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής για το κλίμα, εστιαστήκαμε περισσότερο στο κλίμα. Παράλληλα, με αυτή τη Σύνοδο Κορυφή στη Γενική Συνέλευση δεν έχω απάντηση να σα δώσω, αλλά στη Σύνοδο Κορυφή για το κλίμα εστιαστήκαμε ουσιαστικά σε θεματικού τομεί. Ε, γιατί στη φύση, στην κλιματική αλλαγή δεν εστιαστήκαμε στην πολιτική διάσταση των κυρώσεων. Το σχολείο για το υποεθνικό επίπεδο συμφωνώ απόλυτα. Θεωρούμε ότι είναι μια τάση πολλά υποσχόμενη, ειδικότερα μεγάλες χώρες και ομοσπονδιακές χώρες όπου τα κράτη όπου υπάρχουν ανεξάρτητες δικαιοδοσίες και η Καλιφόρνια για παράδειγμα το γεγονό ότι η Καλιφόρνια δεσμεύτηκε ε, για όλα αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικό, ανεξαρτήτω του τι συμβαίνει πολιτικά σε όλη την Αμερική. Εμεί θέλουμε αυτή την εμπειρία τη Καλιφόρνια να την να αντιγραφεί και σε άλλα μέρη του κόσμου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Έχουμε διάφορου που θέλουν να ρωτήσουν διάφορα πράγματα. Κύριο Γκάλερ πρώτο. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσει. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τη γενική εικόνα, αυτό θεωρώ τουλάχιστον εγώ δεδομένο. Οπότε εσείς είστε σε θέση να ε, συντονίζετε ή να δίνετε συγκεκριμένες υποδείξεις μέσω των οποίων η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ε, μπορεί να εφαρμοστεί πιο αποτελεσματικά. Τι εννοώ με αυτό. Αν πας να δεις κάποιες χώρες που έχουν σχετικά χαμηλό επίπεδο δέσμευσης όπου η προσπάθεια για να φτάσει από το 0% στο 50% είναι πολύ μικρή. Ενώ ε, το ίδιο ποσό, αν στην Ευρώπη, πάντα κάνω αυτό το παράδειγμα. Φυσικά μπορούμε να αναβαθμίσουμε την τεχνολογία φίλτρων ώστε να καθαρίζει από το 90% στο 95%, αλλά αυτό το 5% θα είναι ένα 5% αλλά θα κοστίσει τόσο πολύ όσο σε άλλες περιοχές του κόσμου που θα μπορούσαμε να έχουμε βελτιώσει 50%. Οπότε η ερώτησή μου είναι, εσείς είστε σε θέση να προσδιορίσετε πού μπορεί κανείς με το ίδιο ποσό χρημάτων που έχουν ελάχιστη επίδραση σε υψηλά βιομηχανοποιημένες χώρες να κάνει τεράστια διαφορά σε άλλα μέρη του κόσμου και να δημιουργήσει αυτή τη ε, ε, σύνδεση μεταξύ αυτών που έχουν τα χρήματα και που θέλουν να κάνουν κάτι αποτελεσματικό και εκείνων που είναι ε, έτοιμοι να το κάνουν αλλά δεν έχουν τα χρήματα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να συντονίσουμε όλους αυτούς ε, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και μετά, σε σχέση με αυτό, η δεύτερη μου ερώτηση αφορά την Αφρική. Μια χώρα που γνωρίζω πολύ καλά, η Νότια Αφρική. Έχουν ε, πολύ άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας τους. Τα πάντα γίνονται με το κάρβουνο, αλλά υπάρχει ελάχιστη ηλιακή ενέργεια. Ε, αν υπήρχε πολιτική βούληση θα μπορούσαν να παράγουν περισσότερα σε αυτό το κλάδο. Υπάρχει κάποιος τρόπος, ε, κάποιο κίνητρο που μπορούμε να δώσουμε σε μια τέτοια χώρα ή σε άλλες περιφερειακές χώρες ε, στον κλάδο αυτό ώστε να μεταβούν σε νέες μορφές ενέργειας. Ευχαριστώ. Ώστε να βοηθήσουν να καταπολεμηθεί καλύτερα η κλιματική αλλαγή. Ευχαριστούμε, Μιχαήλ Γκάλερ. Ο κύριος Καστάλντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την προσκεκλημένη μας που ήρθε εδώ για αυτή τη συζήτηση. Όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, τα συμπεράσματα του Σάμιτ για το κλίμα, του Συνόδου Κορυφής για το κλίμα, στη Γενική Συνάλευση εξέφρασαν σημαντικές ε, φιλοδοξίες, ε, πολλά λόγια, πολλές δηλώσεις, ε, στόχοι φυσικά επιθυμητοί που μοιραζόμαστε όλοι, αλλά δυστυχώς πέραν της ρητορικής ε, ε, διαρωτάται κανείς ε, κατά πόσο θεωρούμε ότι θα αντιμετωπίσουμε κάποιες συγκεκριμένες υποθέσεις όπως τους μεγάλους ρηπαίνοντες την Κίνα, τη ΣΥΠΑ που ξεχνάνε την πολύπλευρη αντιμετώπιση και δεν έχουν συγκεκριμένα σχέδια για αυτή την κατάσταση που είναι επίγουσα. Δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο. Δεδομένου αυτού και δεδομένου ότι κάποιες άλλες ε, χώρες στην Ευρώπη και εμεί ω Ένωση προσπαθούμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, αναρωτιέμαι, ε, έπεσαν, σβήσαν τους διακόπτες και το summit και πώς θα προχωρήσουμε τώρα. Υπάρχει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα που θα μας οδηγήσει σε μείωση ε, πραγματική των εκπομπών. Τι περιθώρια επέμβασης έχετε εσείς, άλλες ε, πιθανές πρωτοβουλίες θεωρείτε δυνατές ώστε να μπορέσουμε να αναγκάσουμε αυτές τις μεγάλες ε, δυνάμεις ε, που προφανώς όπως είπαν και άλλοι συναδελφοί πριν από μένα εξακολουθούν να υιοθετούν συμπεριφορές εντελώς αντίθετες στις δηλώσεις που έχουν υποστηρίξει δημοσίω. Και θεωρείτε ότι είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μη τι άλλο, να παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο για να υποστηρίξει αυτή τη στρατηγική των ΗΠΑ Δημιουργώντα έτσι κατά κάποιο τρόπο έναν χώρο, ένα τραπέζι συζήτηση όπου πέρα των ε, μεγαλοστομιών να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με συγκεκριμένες δράσεις χωρίς απλά να ε, κάνουμε δηλώσεις προθέσεων. Ευχαριστώ. Grazie. And our final speaker is... Τελευταία ομιλήτρια, Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μουσούγια Είμαι από τη Σκωτία, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και βρίσκομαι εδώ γιατί ήμουν και μέλος αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νέα Υόρκη. Και συναντηθήκαμε και με τον διευθυντή σας, τον κύριο Άντερσον. Παρακαλώ πολύ, ευχαριστήστε τον εκ μέρους μας που μας αφιέρωσε χρόνο. Ήταν πολύ χρήσιμη συζήτηση που είχαμε μαζί του για την σημασία των ε, λύσεων που θα βασίζονται στην φύση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που απομένουν να γίνουν ακόμα για την εφαρμογή των στόχων του Παρισιού, για την υλοποίησή τους. Θα πρέπει να επιταχύνουμε και θα πρέπει να γεφυρώσουμε το κενό ανάμεσα στις ε, μεγαλύτερες απαιτήσει για κλιματική δράση αφενός και στην έλλειψη φιλοδοξίας αφετέρου. Οι μικρότερες οικονομίες, οι μικρότερες χώρες όπως ε, τα νησιά Μάρσαλ και άλλα νησιωτικά κράτη βλέπουμε πολύ μεγαλύτερη ε, δράση, πολύ περισσότερη δράση από τις μεγαλύτερες χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα κλπ. Εμείς στην Σκωτία, για παράδειγμα, περάσαμε νομοθεσία που προβλέπει ότι θα μειώσουμε τις εκπομπές μας κατά 75% μέχρι το 2030 και θα τις μηδενίσουμε μέχρι το 2045. Είναι προφανώς ότι, προφανές ότι η Σκωτία επιταχύνει, αλλά χρειαζόμαστε και οι υπόλοιπε χώρε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού να κάνουν το καθήκον τους. Η ερώτηση είναι ποια, ποιες βλέπετε να είναι οι βασικές προκλήσεις στο μέλλον σε σχέση με την επιτυχία των στόχων της COP25 ε, στη Χιλή και κυρίως της COP26 στη Γλασκόβη, στην δική μου πόλη. Τι πρέπει να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχει εντωμεταξύ συμβεί αρκετή πρόοδος. Τέλος, το 2020 θα είναι χρονιά κλειδί, γιατί έχουν αναλυθεί Συγκεκριμένε ε, διασμεύσει ό,τι αφορά τα εθνικά προγράμματα και τις ε, πολιτικές στρατηγικές. Ε, πού πιστεύετε ότι θα βρισκόμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, οπότε δίνω ξανά το λόγο στην κυρία Μσούγια. Να απαντήσω στις τρεις αυτές ομάδες ερωτήσεων. Σε ό,τι αφορά τον αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Είναι καλή ερώτηση. Θα σας πω καταρχήν μία φράση και μετά θα σας την εξηγήσω. Δεν είναι unisex οι λύσεις. Αυτά που μπορεί να αποτελούν λύση για μία χώρα, για μία περιοχή, μπορεί να μην είναι λύση για κάποια άλλη, για παράδειγμα. Σε ορισμένες από τις βιομηχανικές χώρες, όπως για παράδειγμα την Νότιο Αφρική την οποία αναφέρατε, το θέμα είναι πώς θα μεταβούμε, πώς θα εγκαταλείψουμε τον άνθρακα όταν κάποιες από αυτές τις χώρες έχουν τεράστια αποθέματα άνθρακα. Ε, σε άλλες χώρες το πρόβλημα είναι τα υψηλά ποσοστά φτώχειας. Οπότε εκεί πρέπει να δούμε ποιες είναι οι εναλλακτικέ λύσει έναντι των ορυκτών υδρογοναθράκων. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, να δούμε ποια είναι η συνολική εμπειρία σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, η Ευρώπη έχει πολύ σημαντικέ εμπειρίε ε, για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και θα πρέπει αυτέ τι εμπειρίε να τι μοιραστούμε με τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε. Και δεύτερον, να δούμε τι ε, επιστημονικά στοιχεία έχουμε. Για Παράδειγμα, σε θέματα μόλυνσης θάλασσα από πλαστικά χρειάστηκε να έχουμε συγκεκριμένα επιστημονικά στοιχεία. Και θα πρέπει να ενισχύσουμε και τη σύνδεση μεταξύ αυτών. Δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο τα πλαστικά στους ωκεανούς, αλλά και το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τουρισμό ή τους προϋπολογισμούς του κλάδου υγείας σε διάφορες χώρες. Εκεί όλα αυτά θα πρέπει βέβαια να εφαρμοστούν με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα, αλλά αυτές είναι οι βασικές κατευθυντήρες γραμμές σε όλο τον κόσμο. Τώρα σε ό,τι αφορά την Νότια Αφρική. Θα έλεγα ρητά ότι όπως έβλεγε και ένας παλιότερος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, η πολιτική βούληση υπήρχε, αλλά υπήρχαν και εμπόδια. Καταρχήν ένα πολιτικό εμπόδιο εξαιτία τη φτώχεια χώρα, στη χώρα και δεύτερον ε, η μετάβαση από τον άνθρακα ε, σε μια πράσινη οικονομία εμποδιζόταν ή εμποδίζεται από την ανυπαρξία αντίστοιχων ανταγωνιστικών λύσεων σε ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην συγκεκριμένη χώρα. Μετά, τι μπορεί να γίνει για τους μεγάλους μολυντές. Εσείς τι μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να πρώτον να προωθήσετε την πολυμέρεια, την πολυμερή προσέγγιση. Η κλιματική αλλαγή δεν έχει γεωγραφικά σύνορα, οπότε όσο πιο πολύ δρούμε μαζί, με δική σας ηγετική θέση σε αυτό, τόσο το καλύτερο. Η στήριξη των πολυμερών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ, είναι πολύ σημαντική. Αυτό θα περιμέναμε από εσά. Ήδη έχουμε πολύ στενή συνεργασία και μάλιστα έχετε χρηματοδοτήσει και τις δράσεις μας με τα χρήματα των φορολογουμένων σας. Επίσης, το δίκτυο των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορες χώρες του κόσμου μπορεί να βοηθήσει σε συνεργασία με τις δικές μας υπηρεσίες και Στι επαφές μας με τις κυβερνήσει και σε επαφές μας με διάφορους φορεί τοπικά. Αυτά μπορούν να, μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε την υλοποίηση των δεσμεύσεων που ελήφθησαν. Το σημαντικό όμως είναι να επιταχύνουμε, ο χρόνος πιέζει και μειώνεται. Ευχαριστώ πολύ τη συνάδελφό από την Σκοτία. Ε, θα ε, δώσω τα χαιρετίσματά σας στην Ίγκα. Σχετικά με την Συμφωνία του Παρισιού, αυτό που βλέπουμε ακόμα και στις μικρότερες των χωρών είναι να γίνεται κάτι, κάτι να κινείται. Οι, οι, σχεδόν όλες οι χώρες στην Αφρική έχουν εθνικά προγράμματα, για παράδειγμα. Το θέμα είναι να υλοποιηθούν. Αλλά και εμείς θα τις βοηθήσουμε οικονομικά με όποιο τρόπο μπορούμε, έτσι ώστε να τηρήσουν τους στόχους του Παρισιού. Οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη επίση μπορούν να βοηθήσουν. Το 2020 θα είναι κρίσιμη χρονιά. Θα είναι η χρονιά της φύσης, όπως είπε η Ίγκα, και είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Είναι σημαντικό η στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης να ενταχθούν στα εθνικά προγράμματα δράσης. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιο άλλο ερώτημα να υπάρχει από δική σας πλευρά, ούτε σχόλιο. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω θερμά κυρία Τζόης Εμσούγια. Νομίζω ότι η επίσκεψή σας σημειώνεται σε μια πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία, σε μια πολύ επίκαιρη στιγμή. Μετά τις εξελίξεις στη Νέα Υόρκη θα συνεχίσετε το έργο σας με τη δέωσα προσοχή και ε, σίγουρα θα προχωρήσουν όλα αυτά τα θέματα στο πλαίσιο των ΗΠΑ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Εκτιμώ ιδιαίτερα την ευκαιρία που μου δώσατε να ε, συναντηθώ μαζί σας. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, να σας ενημερώσω ότι το επόμενο σημείο θα εξεταστεί και κλεισμένων των θυρών. Επομένως, όσοι δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν, θα ήθελα να τους παρακαλέσω να αποχωρήσουν από την αίθουσα αυτή τη στιγμή.